ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο όλο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Γιώργη Σολέη ο εισηγητής και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω μια δήλωση που έχει ετοιμάσει ο συγητής. Ε, δυστυχώς κολλιέται. Ε, όπως ξέρετε γίνονται κάτι πραγματάκια τώρα στην Ισπανία και κολλιέται. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, συντάσσουμε μια έκθεση, προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα πράγματα σε μια σελίδα. Δυστυχώς βέβαια δεν μπορούμε έτσι να αναλύσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Ανέφερα όμως κάποια σημεία τα οποία είναι τα εξή. Το πρώτο είναι ότι η ενσωμάταση της διάστασης ε, του φύλου ως βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στις εξωτερικές σχέσεις. Η ενίσχυση του Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με ειδικό προϋπολογισμό. Η παροχή στήριξης ε, στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικών ηγετών για να προωθήσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα της 61ης Συνόδου της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών θα περιληφθούν στην πολιτική της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και θα αναφέρουν τις σημαντικές συνεισφορές των γυναικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την δίκαιη κοινωνία. Οπότε νομίζω ταιριάζει αυτό με τη σημερινή συζήτηση, να αυξήσουμε τις προσπάθειες να υλοποιηθούν τα δικαιώματα των γυναικών και να έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης με ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των αυτοκτόνων. Να περιληφθεί επίσης η εκπαίδευση στον πυρήνα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, λαμβάνοντας ιδιαίτερος υπόψη την εκπαίδευση χωρίς κινδύνους, να προωθήσουμε τον ρόλο των γυναικών στην ειρήνευση και στον κοινωνικό διάλογο, ειδικά όταν μιλάμε για την πρόληψη των συγκρούσεων, να καταδικάσουμε κάθε μορφή της βίας ε, κατά των ε, γυναικών και της σεξουαλικής βίας ε, εν πολέμο, την κύρωση της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης σε όλα τις τα μέρη και επίσης μόλις υιοθετήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη έκθεση σχετικά στο Στρασβούργο την εβδομάδα που μας πέρασε. Επίσης σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, προγεννητική φροντίδα, μείωση της παιδικής θνησιμότητας, καθώς επίσης και οικογενειακός προγραμματισμός και εκτρώσεις. Αυτά μπορούσε να πει δηλαδή. Αλλά ήθελε επίσης να αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα και ήθελε επίσης να αναφέρει πρώτα απ' όλα τη συγκεκριμένη κατάσταση μεταναστών και προσφύγων. Το αναφέραμε αυτό πέρσι, αλλά βεβαίω το μιλάμε για τα τρομοκιώματα, πρέπει να ξανααναφέρει και την κατάσταση ΛΟΑΡ κλπ. Και βεβαίω ε, έχουμε όλη αυτή την συζήτηση και νομίζω ότι μπορεί να επεκταθεί και με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω τον λόγο στους και όλες από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Μπιλιάνα Μπορζάν. Η κυρία Μπορζάν όμω επίση κολλιέται λόγω ανηλυμένων υποχρέωσεων στην Κροατία. Θέλει να σας ευχαριστήσει για την εξαιρετική γνωμοδότηση που είναι πολύ ισορροπημένη. Αντιλαμβάνεται ότι ε, υπήρχε ένας περιορισμός ε, στο μήκος και θα υποβάλει τροπολογίες που ελπίζει να υποστηριχθούν. Θα αναφερθεί στο θέμα της βίας ε, της έμφυλης, ε, αναγκαστικούς γάμους, ε, γυναικείο γενετικό ακροτηριασμό και το εμπόριο λευκής σαρκός. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος ε, διακίνηση ανθρωπίνων όντων και ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια γίνονται λιγότερο ανεκτικές. Η Μπιλιάνα θέλει να τονίσει την σημασία του ρόλου των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η Μπιλιάνα επίσης ε, πιστεύει πως η οικονομική ενδυνάμωση είναι ο τρόπος για να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και τον αλφαβητισμό. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, να συνδικαλιστούν και δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στην υγεία. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν δωρεάν παροχή υγείας, ειδικά περιγενετική. Επίση, θα ήθελε η Λιάννα να τονίσει το θέμα της ε, βίας ε, που υφίστανται οι γυναίκες ε, και τα ζητήματα αντισύλληψης και έκφρωσης. Πρέπει επίσης να καταθέσουμε τους νόμους ή την πίεση των κρατών που επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης, ειδικά για γυναίκες και λοιπά φύλλα. Ε, σε κάποιες ε, κατηγορίες επίσης, ε, σε κάποιες χώρες η ομοφιλοφιλία είναι έγκλημα. Η Χιλιάνα θέλει να πει ότι δεν μπορούν οι θρησκευτικέ παραδόσεις να δικαιολογήσουν όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά τη βία εις βάρος των γυναικών και κοριτσιών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να δείξει ότι στηρίζει την ενσωμάτωση του φίλου σε όλες τις δράσεις. Άλλοι βουλευτές. Η Ελεονόρα Φορέντσα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να... Ευχαριστώ και θα πρέπει να την ΚΟΕ βεβαίως, ευχαριστώντας την συγκεντρική και τον εισηγητή για νομίζω ότι όλα αυτά που θέλαμε καλύπτονται στο σχέδιο κειμένο. Θα κατεβάσουμε βέβαια ως κοιόδης συγκεντρία για την ΓΚΟΕ κάποιες τροπολογίες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να ενισχύσουμε τα όσα ήδη ε, λέει το κίνημα. Και ε, τα είπαμε στην τελευταία ολομέλεια για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και των ομοφιλοφίλων κλπ. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δεν αφορούν μόνο κάποιες ε, ομάδες ειδικών συμφερόντων, γι' αυτό και θα κατέβασουμε κάποιες τροπολογίες. Αυτά τα δικαιώματα εκφράζουν με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν επίσης ε, δυσμενείς διακρίσεις, υπάρχει το pay gap, υπάρχουν τα θέματα στην πρόσβαση στην ε, κατάρτιση, υπάρχουν οι πρόοροι γάμοι και υπάρχει πάρα πολύ βία. Άρα θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουμε τις γυναίκες και τους ε, ΛΟΑΔ ε, ούτως ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τα δικαιώματά τους ε, και να απολαύουν επίσης και ασφαλείας. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται τον οικογενειακό προγραμματισμό, θα πρέπει να προέρχονται συμβουλές σχετικά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνέπειες για το γυναικείο θέμα ε, των αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν την υπόθεση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει αυτά να γίνουν κατεπηγόντων. Έχουμε τον πέμπτο στόχο του ΟΗΕ ούτω ώστε θα πρέπει να πετύχουμε την ισότητα σαν στόχο του θεματολογίου 2030 στα πλαίσια επίσης των ε, βιώσιμων στόχων ανάπτυξης ή Πρόεδρος. Έχουμε άλλους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι, σας ευχαριστώ και σας ε, υπενθυμίζω ότι οι προθεσμοί για τι τροπολογίες είναι τη Δευτέρα Δεκάτου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 6 Δεκάτου. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε τώρα στο σημείο υπερθυμών 6 που αφορά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων πρωτοβουλία πλευράς των κρατών μελών και έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για να συζητήσουμε. Η υποφαινομένη είναι η συγκεντρία. Συνάδελφοι. Θα σας παρουσιάσω ως συγκεντρία κάποιες σκέψεις μου. Αυτή η πρωτοβουλία είναι βασικό χρηματοοικονομικό μέτρο της Ένωσης. Πρόκειται να βοηθήσει ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Έχει αυξηθεί δραματικά λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. Με αυτή την ε, πρωτοβουλία <clears throat> θα καλυφθούμε με διάφορα προγράμματα ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους άνεργους νέους. Αυτούς που δεν έχουν καταγραφεί ως άνεργοι ούτε έχουν μπει στην επαγγελματική κατάρτιση. Έχουμε μείωση από το 13 πάντως όσον αφορά τη αριθμού των εργωνίων στο 13. Από το 13 Και αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι η μόνη που έχει βοηθήσει στην υπόθεση. Αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί, θα πρέπει να αξιολογηθεί γιατί έχει συμβάλει στις καλές εξελίξεις. Πάντω, τα καθημερινά μα έχουν δώσει πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά στοιχεία όσον αφορά την υποβουλία να απασχολήσει των νέων, ιδίω όσον αφορά τον αντίκτυπο στου νέου και στι νέε. Πάντω γνωρίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία απασχόληση των νέων παρέχει ευκαιρίε. Ευκαιρίε που 48% ανδρών και πενταδίσκων των γυναικών τι έχουν εκμεταλλευτεί. Πολύ θετικό αυτό, διότι έτσι φαίνεται πως η πρωτοβουλία αποδίδει αποτελέσματα και ότι είναι μια προσέγγιση στοχευμένη. Έτσι γίνεται αρρωγή εξατομικευμένη. Πάντως, έχουμε μια σειρά διαφορετικών και συγκεκριμένων λόγων γιατί δεν βρίσκουν δουλειά είναι πολλές φορές. Οι νεαροί και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες ε, έχουν μικρά παιδιά, έχουν διάφορες φροντίδες όσον αφορά το σπιτικό τους και πολλές φορές θέλουν να καταρτιστούν καλύτερα. Όμως Λόγω αυτών όλων των υποχρεώσεών τους δεν μπορούν να σταδιοδρομήσουν με τρόπο πιο αξιόλογο. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Είναι σημαντικό πως τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας θα πρέπει λίγο να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Θα πρέπει να οργανωθούν καλύτερα για να δουν ποιε είναι οι επιπτώσεις, να γίνουν σχετικέ μελέτε και έτσι να είναι καλύτερη η στόχευση αυτή της πρωτοβουλία. Να βρεθούν οι κατάλληλες μέθοδοι, ούτω ώστε να καλύψουμε νεαρούς άνδρες αλλά και γυναίκες που δεν έχουν σπουδάσει και δεν βρίσκουν δουλειά γιατί έχουν ένα σωρό φραγμούς και εντοπίζουν και δεσμένες διακρίσεις. Αν θα πρέπει να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να βγουν από την αγροεργασία να μπορούν να επανέλθουν. Αυτό να ισχύσει και για την ένταξή τους και πάλι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, να υπάρξουν υπηρεσίες, ε, αρρωγή όσον αφορά το μεγάλωμα των παιδιών, όσον αφορά την υποστήριξη των ε, ε ηλικιωμένων, οπότε σε όλους τους κλάδους της ε, οικονομίας και σε επιστήμη, ε, σε επιστήμη παντού, να βοηθήσουμε τις ε, γυναίκες και τις νεαρές γυναίκες να μπορέσουν να βρουν τη θέση τους εκεί. Πάντως παρά την πρώτα που έχει σημειωθεί, ακόμα υπάρχουν υψηλά ποσοστά ενεργεία σε κάποια κρατημέλη. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την πορεία της υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Να υπάρξει σωστή προοικοδότηση στα πλαίσια της περιοδισχύως του πολιετούς ημισονομικού πλαισίου. Να δοθούν κίνητρα, ούτω ώστε να μπορέσουν αυτές οι γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτά ήθελα να σας πω με συντομία για το σχέδιο ε, κειμένου μου. Σας ευχαριστώ για τις συνεργασίες και τώρα να δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδες ηγητές. Και πρώτα πρώτα η κυρία Πέτυρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να επισημάνω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε και να βρούμε επαρκείς ε, λύσεις. Ε, τα κονδύλια που πηγαίνουν σε αυτήν την πρωτοβουλία και για εγγυήσεις ακόμα δεν έχουν δώσει κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολο για τους νέους να βρουν μια μόνιμη θέση εργασίας και να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία. Και πρέπει να πω ότι στην Κροατία 20.000 νέοι έφυγαν ε, αναζητώντας εργασία κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες ολόκληρης της Ευρώπης ε, και πρέπει ακριβώ να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για να προσαρμοστούμε στην αγορά του κάθε κράτους μέλους. Και πρέπει οπωσδήποτε οι νέοι να εμπλακούν περισσότερο και καλωσορίζω τις λύσεις που προτείνεται γιατί αφορούν ακριβώς την εφαρμογή των πτυχών εκείνων ε, που δεν έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερος συντονισμός στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μόνο μέσω τέτοιας ε, συνεργασίας και συντονισμού πολιτικών και χρηματοδότησης ε, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Δηλαδή, οι θέσεις εργασίας για τους νέους. Θα πρέπει επίσης να στοχεύσουμε σε ομάδες ε, ναι, χαμηλότερη εκπαίδευση και βεβαίως ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς ε, που δεν κατάφεραν ακριβώς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και έχουμε βέβαια και το θέμα των περιοχών της υπαίθρου. Είναι δύσκολο να ρυθμιστεί το θέμα της απασχόλησης, ειδικά αν μιλάμε για οικογενειακά ακροκτήματα και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι δυσκολότερο για τις νεαρές γυναίκες να βρουν δουλειά από ό,τι για τους άντρες. Και πρέπει επίσης να δώσουμε βάρος σε αυτό στην έκθεση και στο πλαίσιο του και εμείς έτσι θα διατυπώσουμε τις ε, τροπολογίες μας. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο τώρα στην κυρία Χουσμένοβα από την Άλντε. Σε ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε σας γιατί βεβαίως εργαστήκατε σκληρά για την έκθεση αυτή. Όπως είπατε, η πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση των νέων δημιουργήθηκε για να βοηθήσουμε τους ανεργούς νέους. Και το σκεπτικό ήταν να δώσουμε οικονομική στήριξη σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερος υψηλή η ενεργεία των νέων και με αυτόν τον τρόπο θα έχουν εκείνη προτεραιότητα της ε, πολιτικής της Ένωσης. Οπωσδήποτε συμφωνώ με την γνώμη της εισηγήτριας ότι έχει κρίσιμη ε, σημασία να εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε διαφάνεια στο πώς α, ε, διατίθενται αυτά τα κονδύλια. Πρέπει να έχουμε τις σχετικές εγγυήσεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και βεβαίως ε, μέχρι το 2080 θα έχουμε δύο εργαζόμενους ανά έναν συνταξιούχο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους νέους στην αγορά εργασίας. Και οπωσδήποτε εγώ σας συγχαίρω για την επιτυχία της πρωτοβουλία για την απασχόληση της νεολαίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σημαντικό είναι βεβαίω να μιλήσουμε και για την ισότητα και για την ενεργό συμμετοχή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Πούνεβα. Σκέψεις τι ήταν να μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Την Πέμπτη επιστρέψαμε από την αποστολή που διοργάνωσε με αφορμή τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης για την πρωτοβουλία για την νεολαία Επιτροπή Απασχόληση και Οικονομικών Υποθέσεων στη Σλοβενία και την Κροατία. Τα μαθήματα που πήραμε ήταν πολλά και από τις δύο από αυτές χώρες, μια πρόσφατα ενταγμένη και μια για χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, όμως θέλω να μοιραστώ μαζί στην ουσία τη επίσκεψη αυτής. Η επένδυση στην νεολαία είναι επένδυση στο μέλλον των παιδιών μα και το δικό μας. Πριν φτάσουμε όμως στην επένδυση αυτή, πρέπει να θέσουμε μερικά ερωτήματα στον εαυτό μας. Πώς όμως θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων που μετά από σχεδόν μια δεκαετία κρίσης το ποσοστό της παραμένει απαράδεκτα υψηλό. Πώς θα διασφαλίσουμε τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη στο δημόσιο και την ανάπτυξη, όπως δήλωσε πριν μερικές μέρες ο κύριος Δράγκη από το Τουβλίνο. Ο ίδιος φρόντιζε να μας επιθυμίσει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αλλά ξέχασε να μας πει το πιο σημαντικό, ό,τι ανασυμβεί ή το παραπάνω, αυτά που ουσιαστικά πρέπει να επιδιώξει Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εργαλειοποίηση των νέων στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της, της προηγικότητας. Πώς μπορούμε ακόμα να μιλάμε για καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ακόμα επιτρέπουμε να υπάρχουν συμβόλαια δυνικών ορών πώς μπορούμε να συγχαίρουμε την Επιτροπή που αποφάσισε να ρίξει μερικά ακόμα ψύχολα στην πρωτοβουλία για την νεολαία, ενώ ζητά επιπλέον περικοπές σε μισθούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές πώς περιμένουμε να εφαρμοστεί ουσιαστικά η εγγύηση για την νεολαία και για τις νέες γυναίκες εργαζόμενες όταν ακόμα δεν έχουμε λύσει στοιχειώδη θέματα όπως την άδεια μητρότητας και τις γονικές άδειες. Πώς οι νέες γυναίκες με αναπηρία θα βγουν στην αγορά εργασίας όταν το εργασιακό περιβάλλον δεν είναι προσβάσιμο. Τι θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι για μια άλλη φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα λάθη των πολιτικών του παρελθόντος οι οποίοι κρατούν έρημες στις πολιτικές του μέλλοντος. Δεν τα κοραστώ να το λέω, χωρίς ένα θέλος στο ντόγμα της πολιτικής που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική λιτότητα, αυτές οι πολιτικές δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ρίχνουν νερό στο μήλο της φτώχειας και της ανεργίας. Πριν μερικές εβδομάδες, στην Επιτροπή Απασχόληση ήρθε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση η πρωτοβολία της αναπληρώτριας Υπουργού πολέμησης της Αναργίας της Ράνιας Δονοπούλου. Ανάμεσα σε άλλα πρότεινε την εξαίρεση από το υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος μέρος των κοντιλιών που διατίθεται για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς η παρέμβαση για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασία συνιστούν επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή είναι μια πρόταση που οφείλουμε να στηρίξουμε όλοι μας. Τέτοιες πρωτοβολίες χρειαζόμαστε στην Ευρώπη αν θέλουμε να δούμε τα ποσοστά της ανεργίας να πέφτουν και σοβαρές επενδύσεις σε σταθερές θέσεις εργασίας να γίνονται. Η γνωμοδότηση της συνάδελφου Μπλίνκεβιτσιούτη είναι σε καλό δρόμο και είμαι σίγουρη πως στο τέλος μαζί και με τις τροπολογίες θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο να καταθέσουμε. Νομίζω πως με τις τοποθετήσεις μου έχετε ήδη καταλάβει που θα δώσω έμφαση για τη δική μου πλευρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα. Κυρία Ρέτγε, έχετε το λόγο. Όχι, πρώτα να μην επαναλάβω όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι, αλλά να σας ευχαριστήσω και εγώ για το σχέδιο κειμένου που νομίζω ότι μας πάει στη σωστή κατεύθυνση για την πρωτοβουλία. Ήδη έχει αποδώσει καρφούς ταυτόχρονα, όμως Χρειαζόμαστε περισσότερες ε, κινήσεις για να το πολεμήσουμε την ανεργία. Μπορεί τα νούμερα να είναι κάπως πιο ρόδινα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές, αλλιώς οι νέοι που έχουν τόσο ευάλωτες θέσεις απασχόλησης ή που δεν έχουν δουλειά να θεωρήσουν ότι μια, μια που τα στατιστικά πάνε λίγο καλύτερα δεν δίνουμε δεκάρα για αυτούς. Πάντως θέλω να σας πω ε, άλλα δύο θέματάκια θα πρέπει στο κείμενο να αναδείξουμε κάπως περισσότερο αυτό το οποίο λέτε ότι χρειάζεται κάποιο πιο εξοδομικημένη προσέγγιση έτσι να φέρουμε τον ε, κόσμο πιο όντα με, περισσότερες περισσότερε προοπτικές προοπτικέ, όσον αφορά του μακρόχρονου ανέργου δηλαδή, να έχουμε προγράμματα στοχευμένα, ιδιαίτερος, ιδιαίτερο στοχευμένα για τις γυναίκες όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Οι γυναίκες πολύ συχνά έχουν πάρα πολλές ε, ευθύνες φροντίδας και ε, έχουν το θέμα των παιδιών τους. Αυτό να ληφθεί υπόψη. We are um, planning these programs and see how we can individually... Θα δούμε πώς το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει με εξατομικευμένο τρόπο και έτσι να μπουν ξανά στα ώρα αυτές οι γυναίκες. Επίσης, ε, έχουμε κάποιες μικρές ελλείψεις στο κείμενο, ιδίω όσον αφορά τα στερεότυπα που πρέπει να γκρεμίσουμε, Πρόεδρε, όπω και εσεί αναφέρετε, είναι σημαντικό επομένω για τα μέτρα που αφορά τι δεξιότητε και την κατάρτιση. Σε αυτά τα προγράμματα κάτι να προτείνουμε. Και να μην λέμε ότι τα αγόρια γίνονται μηχανικοί και οι γυναίκε κάτι άλλο. Τέλο πάντων, οι γυναίκε ότι πάνε στις υπηρεσίε φροντίδας δηλαδή μόνο. Άρα να δούμε τι γίνεται γενικότερα για κάθε απασχόληση. Έτσι θα γίνει αξιόλογη η γνωμοδότηση όπως και πιστεύω ότι θα είναι και ευχαριστώ για τη συζήτηση. Η Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ρέντ και θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Mm. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Σα ενημερώνω ότι οι προθεσμοί της τροπολογίας είναι η Δευτέρα Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε στις 6 Νοεμβρίου. Οπότε και θα έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Εγώ, ως ε, συντάκτης, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συγητές, να τους ευχαριστήσω για παρατηρήσεις, για σχόλια, και στο μέλλον να συνεργαστούμε. Έχουμε κοινό στόχο να καλύψουμε νέους και νέες. Θα πρέπει να μπορούν να βρουν απασχόληση ποιότητας. Προχωρούμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7. Όσον αφορά την ε, αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό, προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων. Α, μισό λεπτό. Πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Μονόλεπτο. Ένα λεφτάκι. colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά καλώς, σας καλωσορίζω σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Και την ε, ευημερία των γυναικών. Έτσι οι γυναίκε και οι οικογένειε θα μπορέσουν να προγραμματίσουν καλύτερα το μέλλον του, θα υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Αύριο, 26 Σεπτεμβρίου, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα της σύλληψης και επί τη ευκαιρία η Επιτροπή Γυναικών αποφάσισε να οργανώσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων ως ευκαιρία για να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Γιάνν Πάχλερ επικεφαλής ε, της αρμόδιας διεύθυνσης στην ε, ΔΕΒΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μας καλέσατε εδώ και βεβαίως ε, είναι πάντα μεγάλη ευκαιρία να μιλάμε για την οικογενειακό προγραμματισμό, κάτι το οποίο ωφελεί πολλούς τομείς αγαπητούς εμάς. Είναι γνωστό ότι μειώνει τους κινδύνους, τους σχετικούς με την κοιμοσύνη, μειώνει την ανάγκη έκτρωσης, ε, την παιδική θνησιμότητα και τα αφροδίσια μεταξύ των οποίων και το HIV-AIDS ε, και για και για τα παιδιά μειώνει τις ε, εγκυμοσύνες ανηλίκων οπότε τα κορίτσια μαθαίνουν περισσότερα γράμματα και μπορούν μετά να δουλέψουν και έτσι επιβραδύνεται η ανάπτυξη του πληθυσμού και τέλος μπορούν οι γυναίκες να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, που αφορούν τι να αποφασίζουν μόνες τους για αυτά τα θέματα. Έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση που θα είναι αποτελεσματική και θα βασίζεται σε στοιχεία και θα έχει και πολύ καλή οικονομική απόδοση είτε από την πλευρά της υγείας, του φίλου ή από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναρωτιόμαστε γιατί ε, Ακριβώ η παρέμβαση αυτή δεν διατίθεται σε κάθε γυναίκα που την χρειάζεται. Αυτό ισχύει ειδικά στην Αφρική όπου μόνο 20-30% των γυναικών ε, έχουν πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό που θα ήθελαν. Σαφώς λοιπόν έχουμε μια πρόκληση εδώ πέρα ειδικά για τις χώρες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να διαθέσουν αυτές οι υπηρεσίες στον πληθυσμό και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό σε αυτές τις χώρες. Προσπαθούμε να υπάρχει καθολική παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι ίδιες αξίες που έχουμε για τα δικά μας συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να ισχύουν και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό σημαίνει να ερχόμαστε σε επαφή με τις ε, ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια, να τις στηρίζουμε μέσω παρεμβάσεων που βασίζονται σε στοιχεία, σώζει ζωές και αυξάνει την ευμερία. Η δέσμευση της Ένωσης για την ισότητα των δύο αφορά βεβαίως ε, και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών ε, και αναφέρεται και στο, στη νέα συνένεση της Ένωσης για την Ανάπτυξη που ενέκρινε τον Ιούνιο Συμβούλιο Κοινοβούλιο και Κομισιόν και έχουμε και το σχέδιο δράσης 2016-2020 ε, που ενέκρινε το Συμβούλιο το Σεπτέμβριο 2015 επιπλέον η προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, είναι θεμελίως λήθος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα υγείας στο τωρινό ΠΔΠ 2014 2020 τα μισά από αυτά σε διμερεί προγράμματα υγείας σε 17 χώρες κλειδιά και τα άλλα μισά μέσω παγκοσμίων πρωτοβουλειών όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, φυματίωσης και ελονοσίας, ε, την Παγκόσμια Συμμαχία για τα εμβόλια και το πρόγραμμα τροφίμων του ΙΕ. 230 με 240 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται κάθε χρόνο σε προγράμματα που αφορούν την απαραγωγική υγεία και την υγεία νεογνών και παιδιών. Από αυτά 40 με 45 εκατομμύρια κάθε χρόνο πάνε συγκεκριμένα για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Νωρίτερα φέτος λοιπόν ε, είδαμε πως η νέα Αμερικανική κυβέρνηση επανέφερε τη λεγόμενη πολιτική του Mexico City με στόχο να κόψει την διεθνή χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων. Επίτροπος Νίμιτσα είπε πως ανησυχεί ιδιαιτέρως για την επαναφορά αυτής της πολιτικής και το τι σημαίνει αυτό για ευάλωτα κορίτσια και γυναίκες για τις υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού. Κινδυνεύουμε εδώ πέρα η πρόοδος της τελευταίας δεκαετίας για τα δικαιώματα των γυναικών να πάει χαμένη. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την απόφαση να μηδενιστεί η διεθνής βοήθεια, ε, κατά το οποίο από ό,τι φαίνεται θα οδηγήσει στην έγκριση ενός νόμου από την αρμόδια υποεπιτροπή με ένα πλαφόν 120 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι πολλά λεφτά αλλά ακόμα σημαίνει ότι υπολείπονται κατά πολύ από τα 605 ε, εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται. Οι καλεσμένοι μας εδώ πέρα θα μας εξηγήσουν το τι σημαίνει αυτή η περικοπή η ΕΠΑ είναι και θα παραμείνει σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική, αλλά ο Επίτροπος Νίμιτσα είπε ότι δεν θα ήθελε η ευρωπαϊκή πολιτική να ακολουθεί τα όσα κάνουν ή σταματούν να κάνουν οι άλλοι. Αυτό είπε πως πρόκειται για ε, να συνέδριο υπέρ των γυναικών. Είναι γνωστό πως η ανάπτυξη και οι γυναίκες είναι πρώτη του προτεραιότητα. Και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών σε τέτοιες υπηρεσίες ανά τον κόσμο και μαζί με τους εταίρους μας Παγκοσμίω θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα για να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους και τελικά την υγεία τους. Και σκοπεύουμε να πείσουμε και τις κυβερνήσεις να ξοδέψουν εθνικούς πόρους ε, σε τέτοιες υπέροχες παρεμβάσεις και να καταστήσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό ε, διαθέσιμο σε όλους. Τα δικαιώματα αυτά είναι βασικό τμήμα των δεσμεύσεων για την ισότητα, όπως αναφέρεται στο σχετικό σχέδιο δράσης. Ο Επίτροπος Νίμιτσα το ανέφερε αυτό στην διάσκεψη c Decides όπου μιλήσαμε για κλιμάκωση και καλύτερη πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Πρώτη μας ε, έκθεση λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ ξεκίνησαν μια νέα συνεργασία για να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με ένα ξεχωριστό προπολογισμό μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία που θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε μια στρατηγική συνεργασία με τον ΟΗΕ για να επιβεβαιώσουμε την απαρασάλευτη ε, δέσμευσή μας για την ενδυνάμωση των γυναικών. Σημαντικό κομμάτι των 500 εκατομμυρίων θα πάει και σε ένα πιστεύουμε, στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλες εταιρείε. Επίσης, εξετάζουμε και άλλες επιλογές πιο στοχευμένες στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του πολιετούς προγραμματισμού. Οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει περιλαμβάνουν 100 εκατομμύρια ευρώ για την ισότητα των φίλων και δικαιώματα των κοριτσιών για την περίοδο 2014-2020 και 18 δισεκατομμύρια έχουν ήδη δεσμευτεί. 20 εκατομμύρια σε προμήθειες του προγράμματος τροφίμων του ΟΗΕ για να βελτιωθεί η ζήτηση για και η πρόσβαση σε είδη ε, οικογενειακού προγραμματισμού και 30 εκατομμύρια ευρώ για να ζητήσουμε πρόσφορες ε, για την πρόθεση της ισότητας και την ενδυνάμωση των γυναικών. Κατ' ουσίαν δεν ε, γεμίζουμε εμείς το κοινό που άφησαν άλλοι, αλλά επενδύουμε στρατηγικά το χρήμα των προλογουμένων εκεί όπου θα έχουμε μεγάλη απόδοση όταν μιλάμε για ζωές που σώζονται και για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύεται στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάτλερ για την τοποθέτησή σας. Η κυρία Στάινακερ λαμβάνει τον λόγο του τμήματος ε, των Βρυξελών του Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα ένα σύντομο βίντεο το οποίο ε, μας δείχνει παράδειγμα από την χώρα Μπενίν για το πώς μπορεί να κάνει κανείς οικογενειακό σχεδιασμό στην πράξη και υπό δυσχερείς συνθήκες. Καμιά φορά χρειάζεται να είναι κανείς και κάπως δημιουργικός και να κάνει και μια έξτρα προσπάθεια. Ορίστε λοιπόν.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 Να λοιπόν αυτό ήταν ένα παράδειγμα ε, του πώς μπορούμε να προσφέρουμε ε, ε, οικογενειακό σχεδιασμό κάνοντας μια έξτρα προσπάθεια ε, δηλαδή πηγαίνοντας κάπως παραπέρα όπως λέμε στα αγγλικά. Να επανέλθουμε όμως για λίγα λεπτά. Α, ωραία, λειτουργεί καλά το σύστημα με τη διαφάνεια. Σας επανέλθουμε στο γιατί είναι τόσο σημαντικός ο οικογενειακός σχεδιασμός. Είναι σημαντικός διότι δίνει τη δυνατότητα, δίνει την ε, δύναμη να χρησιμοποιήσει το αντισυλληπτικό γυναίκα εάν θεωρήσει ότι χρειάζεται. Και είναι και στο ανθρώπινο δικαίωμα. Διότι, διότι ο οικογενειακός σχεδιασμός σώζει ζωές. Αποφεύγουν τα αντισυλληπτικά, δηλαδή βοηθούν να αποφευθούν ε, ανεπιθύμητες ε, και που ενδεχομένως μπορεί να έχουν και προβλήματα στη διάρκεια της ε, κύσεως Μειώνουν λοιπόν ε, σημαντικά και τους κινδύνους για τις μητέρες αλλά και για τα νεογέννητα. 240 εκατομμύρια γυναίκες και νεαρά κορίτσια που δεν θέλουν να μείνουν έγκυες όμως δεν χρησιμοποιούν σύγχρονα συλληπτικά είτε διότι δεν έχουν τα μέσα να τα αγοράσουν είτε διότι δεν γνωρίζουν είτε διότι δεν έχουν πρόσβαση ναι. στις κλινικές, είτε διότι αντιμετωπίζουν την καταδίκη της κοινωνίας και το στίγμα. Δεύτερο, ο υπενεκός σχεδιασμός δίνει δύναμη στις γυναίκες και στα κορίτσια, διότι είναι ουσιώδης για την επιτυχία, για την επίτευξη μάλλον, της ισότητας των ευκαιριών, διότι η γυναίκα τότε αποφασίζει πότε θα αποκτήσει παιδιά. Μπορεί έτσι να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της. Αυξάνει η αυτονομία της μέσα στο νοικοκυριό και η δύναμή της. Αυτό προσφέρει στη γυναίκα οικονομική ασφάλεια, ευημερία, βεβαίως και στις οικογένειες. Τρίτο, ο οικογενειακός σχεδιασμός, το είπε κάποιος πριν αυτό, είναι σημαντικός και για την παγκόσμια οικονομία και τελικώς είναι και ευθυνός τρόπος εάν ε, λάβει κανείς υπόψη τα, ε, τα ωφέλη που ε, αποδίδει. Για κάθε ε, ευρώ ή κάθε δολάριο που δαπανούν ε, στον οικογενειακό σχεδιασμό εξοικονομούν 5 δολάρια από άλλες φροντίδες υγείας κλπ. Η, συνολική πρόσβαση στις φροντίδες υγεία που περιλαμβάνουν και τον οικογενειακό συνδυασμό αποδίδει αξία της τάξης του 120 δολαρίων για κάθε δολάριο που επενδύεται. Ένα δολάριο επενδύει 120 ε, λαμβάνεις πίσω. Εποφελούνται από την σύγχρονη αντισύλληψη που εκτός του ότι εξασφαλίζει ένα θεμελιώδης ανθρώπινο δικαίωμα, αποφεύγονται και 76.000 θάνατοι ε, των ε, ε, γυναικών κατά τον τοκετό. Και βεβαίω αποφεύγονται και πάρα πολλές ανεπιθύμητες σκήσεις. σημαντική, όπως είπα, απόδοση της επένδυσης, ας το πω έτσι. Τώρα, πώς προσφέρουμε συνολικό οικογενειακό σχεδιασμό. Θα θυμάστε ότι το 2012 στη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής για τον οικογενειακό σχεδιασμό, σε εκείνη την πολύ σημαντική διάσκεψη, είχε αναλυθεί η δέσμευση, ο στόχος δηλαδή, μέχρι το 2020 να προσφερθούν σε 120 πρόσθετα εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια που δεν έχουν πρόσβαση στον οικογενειακό σχεδιασμό, να τους προσφερθεί πρόσβαση στην αντισύλληψη. Στις 12 Ιουλίου φέτος έγινε άλλη μια διάσκεψη για τον οικογενειακό σχεδιασμό για να καταγραφεί η πρόοδος που έχει συμβεί σύμφωνα με τους στόχους του 2020. Και υπάρχει πρόοδος. Μέσα σε τέσσερα μόνο χρόνια έχουμε μπορέσει να προσφέρουμε οικογενειακό σχεδιασμό σε 32 εκατομμύρια περισσότερα ε, κορίτσια και γυναίκες. 300 εκατομμύρια γυναίκες που χρησιμοποιούν σύγχρονα τα συλληπτικά χάρη στο πρόγραμμα αυτό στην Ανατολική και Νότια Μεσημβρινή δηλαδή Αφρική πάνω από 20% των κοριτσιών και γυναικών χρησιμοποιούν σύγχρονες ε, μεθόδους αντισύλληψης. Δεν μπορείτε να διαβάσετε μικρά γράμματα διαφάνειας, θα σας λέω εγώ. Λοιπόν, στη Δυτική Αφρική, όπου πάντοτε χρησιμοποιούσαν λίγα αντισυλληπτικά, στην Ουαγκαντουγκού, έχουμε ήδη ξεπεράσει τον στόχο του 2015 και κοντεύουμε να φτάσουμε τώρα 2,2 πρόσθετες, εκατομμύρια δηλαδή, πρόσθετες χρήστριες. Έχει γίνει λοιπόν σημαντική πρόοδος, παραμένουν όμως κενά και ιδίω για τις ανήλικες. Το 2016 19,2 εκατομμύρια ανήλικα κορίτσια που είχαμε δεσμευθεί να καλύψουμε στη διάσκεψη του 2012 και εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην οικογενειακό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε, πρέπει να επιταχυνθεί η πρόοδο. Και έρχομαι τώρα στο πρόγραμμα του UNFPA. Πάντοτε σε σύγκριση με τον στόχο του 2020 και βέβαια τους στόχους της ε, ε, αηφόρου ανάπτυξη κλπ. Να λοιπόν βλέπετε στου χάρτες αυτούς τις χώρες όπου προσφέρει η UNFPA υποστήριξη, ιδίω στην υποσαχάρια Αφρική, λίγο στη Λατινική Αμερική και λίγο στην Ασία. 46 χώρες χαμηλού εισοδήματο συνολικά. Χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά θανάτων στη διάρκεια του τοκετού και σημαντικές ανάγκες οικογενειακού σχεδιασμού. Η NFPA είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ε, δωρεάν αντισυλληπτικών. Μια στιγμή όπως είπα είναι το μεγαλύτερο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών προσφέρει την υποστήριξη αυτή. Όπως είπε προηγουμένως ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ΔΕΦΚΟ ε, είναι σημαντική δωρήτρια για το Ηνωμένο Έθνη μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις κάτω χώρες, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, από τις ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή, αλλά και τον Καναδά. Το Ταμείο έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο αμερικανικά δολάρια από τότε που δημιουργήθηκε. Η UNFPA προσφέρει πάνω από το 40% των δωρεάν αντισυλληπτικών σε όλο τον κόσμο και φτάνει στα χέρια 20 εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών. Προσφέρει επίσης στήριξη για τους στόχους NFPA και άλλους παγκόσμιους στόχους. Το 1 τρίτο των γυναικών που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά στις 69 χώρες χρησιμοποιούν αγαθά που προσφέρουν η UNFPA. Και είναι κρίσιμο να επιτευθεί η πρόσβαση σε οικογενειακό σχεδιασμό, ιδίω για τους στόχους 3 και 5 που έχουν σχέση με τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία των στόχων της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Η UNFPA προσφέρει και αντισυλληπτικά σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προσφέρουν με τη σειρά τους οικογενειακό σχεδιασμό σε διάφορες χώρε. Όλα αυτά βέβαια σε ό,τι αφορά την προσφορά αγαθών, την προσφορά των ειδών αυτών. Αλλά προσφέρουν και στήριξη για να περάσουν από την φάση στήριξης μεσοδορητών στην, ε, στο να οικειοποιηθούν τις πολιτικές για τον οικογενειακό σχεδιασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, διότι τελικώς από εκεί θα χρειαστεί να βρεθούν τα χρήματα. Τώρα βέβαια πάντα πρέπει να μιλεί κανείς και το κενό, για το κενό χρηματοδότησης. 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω θα κοστίσουν η συνολική κάλυψη. Λέμε εκεί 5 δισεκατομμύρια στη διαφάνεια, στην πραγματικότητα 5,5 δισεκατομμύρια. Η UNFPA αντιμετωπίζει ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για την ε, περίοδο 2017 έως 20 αυτά για να επιτεθούν στόχοι του 2020. Χωρίς όμως τα ίδια αυτά, τα συντριπτικά, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως δωρητές και χώρες προγράμματος. Να έρθουν δηλαδή οι χώρες αυτές και να πληρώσουν το χρηματοδοτικό κενό. Βέβαια, η παροχή και μόνο αντισυλληπτικών δεν αρκεί. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενημέρωση, πληροφόρηση του κοινού, των ε, ανθρώπων, των νέων γυναικών και ανδρών για τις επιλογές που έχουν. Και ιδίω οι νέοι που χρειάζονται πρόσβαση σε ποιοτικό οικογενειακό σχεδιασμό για να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δύναμη να κατευθύνουν τη ζωή τους. Σήμερα, όπως είπα, 240 εκατομμύρια δεν έχουν την πρόσβαση αυτή και χρειάζεται να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι 120 εκατομμύρια πλέον, επιπλέον γυναίκες και κορίτσια. Αυτά είναι από τα πρώτα ορόσημα της πορείας μας, γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι συνολική, παγκόσμια πρόσβαση με το 2030 πλέον ε, σε αντισύλληψη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα το στόχο αυτό. Ο στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένας που να μην έχει πρόσβαση, καμία μάλλον. Και χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων για να μπορέσουμε εν τέλει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την υγεία, αλλά και να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην οικονομική ευημερία και το μέλλον όλων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο των βουλευτών, τι μπορούν να κάνουν δηλαδή οι βουλευτές η πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη για τον οικογενειακό σχεδιασμό έχει σημασία κλειδί για την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών. Τα θέματα αυτά καμιά φορά είναι υπερευαίσθητα ή πολύ περίπλοκα και αποτρέπουν ε, τους ανθρώπους από το να ασχοληθούν, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι αυτό, είναι αυτονόητο. Δηλαδή θα πρέπει πάντοτε να μένει το θέμα αυτό ε, στο θεματολόγιο στην advocacy agenda, ώστε να προβάλλονται τα θέματα του οικογενειακού σχεδιασμού σε κάθε κατάλληλο πλαίσιο. Για παράδειγμα, στη διάσκεψη κορυφή Αφρική Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο, στο High Level Political Forum. Το ίδιο σημαντικό είναι να συνεχιστεί να υπόλογη στι εθνικέ κυβερνήσει για του ε, στόχου SDG, δηλαδή της αηφόρου ανάπτυξης, 3 και 5 και του άλλου βέβαια μα ικανοποιεί η προφορική τροπολογία που ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή σα τη ανάπτυξη για να προσθεθούν 20 εκατομμύρια στον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά για ε, τα θέματα αυτά και ελπίζομαι τελικώ να υλοποιηθεί η δεσμεύση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ιρένη Τρεντία από την από το Διεθνές Δίκτυο ε, Οργανώσεων Γονέων. Ευχαριστώ. Μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα την αντισύλληψη. Μεγάλη ε, και σπουδαία ευκαιρία αυτή για μας. Δύο λόγια για το ακροτήριό σας που ίσως να μην γνωρίζει τον οργανισμό μας που λέγεται IPPF και είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός που ασχολείται με τα ε, αναπαραγωγικά δικαιώματα στον κόσμο. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε τις αλλαγές μέσα από τις οποίες περνούμε και το γεγονός ότι το πολιτικό τοπίο και όχι μόνο το οικονομικό τοπίο έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θαραλέα στάση της και κύριος Επίτροπος Νίμιτσα. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα γενετήσια και αναπαρικά δικαιώματα των γεγονών των γυναικών απειλούνται. Μου ζήτησαν να μιλήσω για την κατάσταση στην Ευρώπη. Ακούσαμε ζητήματα για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, διότι διακινδυνεύεται η πρόοδο που έχουμε επιτύχει. Είναι σημαντικό λοιπόν να ζητήσουμε ή να, να παρακαλέσουμε του ευρωβουλευτέ που είναι παρόντε και παρούσε ότι χρειαζόμαστε και άλλε πολιτικέ υπέρ τη αντισύλληψη, όπω το λέει και η διαφάνεια χρειαζόμαστε και συγκρίσιμες έρευνες ώστε να γίνει σαφές ότι η συνολική πρόσβαση δεν είναι δεδομένη ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθολική πρόσβαση. Διεξάγω μια εκστρατεία η IPPF και που λέγεται I decide, εγώ αποφασίζω. Σας παρακαλώ σκεφτείτε, αναλογιστείτε για λίγα δευτερόλεπτα ποιε είναι οι πιο ευάλωτε ομάδε στην Ευρώπη και στι χώρε σα. Υπάρχουν πολλέ τέτοιε ομάδε. Θα σα έρθουν αυτόματα στο μυαλό ορισμένε, αλλά υπάρχουν και πολλέ άλλε κατηγορίε. Βλέπουμε πολλέ διακρίσει σε βάρο αναπήρων ανθρώπων, ε, κατά νέων και ιδίω ανηλίκων. Πολλά προβλήματα με μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες κατηγορίες και ιδίως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 Και βέβαια, η κατάσταση των μεταναστριών, κυρίως και ιδίως των παράτυπων μεταναστριών και προσφύγων είναι ιδιαίτερα δυσχερής Υπάρχουν φραγμοί όμως και για πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων στην κοινωνία και ελπίζουμε πολύ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για τα πρόσωπα αυτά. Θέλουμε επίσης να επισημάνω στη, σε εσά ότι υπάρχουν και σημαντικές απειλές ε, σε βάρος και όλων των γυναικών στην Ευρώπη. Θα έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει στην Πολωνία για παράδειγμα, διότι ε, έχουν οδηγήσει τα πράγματα αυτά τόσο πολύ κόσμο στη, στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες. Λοιπόν, πολύ, αλλά έγιναν πολλές συζητήσεις για την αντισύλληψη, διότι υπήρχε και σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά ε, με την αντισύλληψη κατεπιουσών καταστάσεων που δίνεται χωρίς συνταγή και αποφάσισε η κυβέρνηση να μην εγκρίνει, μάλλον να μην ε, ε, υπακούσει στην σύσταση αυτή και να μην δώσει την λύση αυτή επιγουσών καταστάσεων σε ορισμένες στις γυναίκες. Ακόμα δηλαδή και θύμα βιασμού στην Πολωνία δεν έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεμελιώδη υπηρεσία, διότι θα πρέπει να βρει γιατρό και φαρμακοποιό που να είναι διατεθειμένοι να τις παράσχουν την ε, κατεπίγουσα αυτή αντισύλληψη. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε απλώς ε, να τα κοιτούμε τα πράγματα αυτά. Βέβαια, παρόλο το ε, σκοτεινό αυτό πανόραμα που σας έδωσα, υπάρχουν και καλά νέα. Γίνονται και καλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στην Γαλλία μέχρι τα 18 οι νέες και οι νέοι έχουν δωρεάν, ε, δωρεάν ιατρική φροντίδα και για τέτοια πράγματα. Και από το 2016 δωρεάν και ανώνυμη αντισύλληψη και ε, ιατρικές συμβουλές δίνονται σε κορίτσια μεταξύ 15 και 18. Στην δε Σουηδία μέχρι και τα 21. Και σε ορισμένα μέρη της χώρας μπορεί να φτάσουν και την ηλικία των 26 ετών. Μεταξύ 21 και 26 έχει η γυναίκα ε, ευθυνότερη πρόσβαση διότι είναι επιδοτούμενες οι υπηρεσίες αυτές. Πάλι, αν σκεφτείτε την κατεπίγουσα αντισύλληψη. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι στη Γαλλία εγκρίθηκε πρόσφατα νέο μέτρο και οι ανήλικες μπορούν να λάβουν την επίγουσα αντισύλληψη όχι μόνο χωρίς συνταγή, αλλά και δωρεάν και απολύτως ανώνυμα. Άρα δεν χρειάζεται καν να δείξουν ταυτότητά τους. Συγκρίνεται τώρα τι κάνει η Πολωνία και άλλες χώρες. Αντιλαμβάνεστε πόσο βαθιές είναι οι διαφορές. Ενώ στη Σουηδία μπορεί να λάβει κανείς την επίγουσα ε, αντισύλληψη σε κάθε ε, κλινική. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στη Γαλλία. Η αντισύλληψη είναι δωρεάν για νεαρές κοπέλες αλλά και για γυναίκες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος. Μπορούν το αυτές να λάβουν ειδική επιδότηση. Έχει δηλαδή δημιουργηθεί ένα σύστημα ενώ στην Πορτογαλία, στον νότο της Ευρώπης, υπάρχει ευρύτατη ε, δωρεάν πρόσβαση για όλες τις γυναίκες. Η Πορτογαλία μάλιστα διατήρησε το μέτρο αυτό και στη διάρκεια των μέτρων λιτότητας. Θα επαναλάβω αυτό που είπε εσεί και διότι συμφωνούμε ότι για το FPA ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πολιτικός πολιτική μάλλον και χρηματοδοτική υποστήριξη για τον οικονομικό σχεδιασμό και από εσά, από το ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Λέει η οργάνωση Mouse Mondial de Femme, η κυρία Σίλβια Λάουσπεργκ, εκπροσωπεί τον οργανισμό αυτό, είναι και αντιπρόεδρος του γαλλόφωνου ε, Συμβουλίου Γυναικών του Βελγίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σας μιλώ εκ μέρους ε, της παγκόσμιας πορείας των γυναικών. Ο σκοπός μας είναι να σταματήσει η βία των γυναικών Έχουμε 6.000 ε, ε, φορείς σε 161 χώρες και σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο διότι η γενικευμένη πρόσβαση στην αντισύλληψη θα πρέπει να αποτελεί τμήμα της πολιτικής ισότητας αλλά και της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών γιατί είναι ε, ότι κατά παράδειγμα τρόπο υπάρχει δυσμένης διάσταση κατά των γυναικών και θα αναγκάζονται λόγω του σώματός τους να γίνονται μητέρες. Όμως πρόκειται περί μεγάλης ευτυχής. Αυτό είναι η μητρότητα. Οπότε έτσι γίνεται κάτι το οποίο κατατρίχει τη γυναίκα ε, σωματικά και φυσικά. Όμως δεν μένει έγκυος η γυναίκα από το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει η ευθύνη που αφορά και την αντισύλληψη. Και οπότε τα θέματα για την έλλειψη αντισύλληψη είναι ακόμα μια ανισότητα τη βάρο τη γυναίκα. Έχουμε κάποιε χώρε όπου υπάρχει οικογενειακό προγραμματισμός, οπότε μια ανεπιθύμητη γη ε, ή άλλοι λόγοι οφείλονται στην έλλειψη τη αντισύλληψη. Οπότε θα πρέπει οι γυναίκε να περιορίσουν αυτή την έλλειψη ελευθερία, θα πρέπει να έχουν τα ενία τη ζωή και του μέλλοντο, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό ε, θα πρέπει να σταματήσει το σαμποτάζ της ε, αντισύλληψης και ξέρετε πόσο φρικτά είναι τα νούμερα τα σχετικά με την εγκατάλειψη των εγγύων, τι γίνεται επίσης με την σεξουαλική βία και τους βιασμούς. Οπότε είναι η αντισύλληψη ένα δικαίωμα, γιατί επομένως θα πρέπει η άμβλωση να είναι ποινικό αδίκημα για πρέπει, γιατί θα πρέπει να προσάγεται με της δικαιοσύνης για αυτό το λόγο, γιατί θα πρέπει να υφίσταται όλες αυτές τις διακρίσεις που καταγγέλλονται από τον ΟΗΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει ε, όχι μόνο στα χαρτιά να έχουν τα ίδια δικαιώματα για όλα, να πρέπει να έχουν και για τον ε, γενετήσιο βίο. Θα πρέπει επίσης να αλλάξει η νοοτροπία, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το να μην μπορεί η γυναίκα να κάνει άμβλωση αποτελεί άσκηση βίας εναντίον τη. Είναι απαράδεκτο ό,τι και να πιστεύει κανεί να δέχεται το μη γυναίκα να έχει κίνδυνο τη ζωή της γιατί δεν μπορεί να κάνει άμβλωση. Και τελικά, ακόμα και στην Ευρώπη, αν κάνουν οι γυναίκες να κάνουν υπό τραγικέ παρόμοιε αμβλώσεις και να πεθαίνουν πολλές φορές αναγκάζονται να μείνουν έγκυες οι γυναίκες ε, πολλές φορές υπάρχει υπάρχουν προβλήματα ορμονικά, υπάρχει παραπληροφόρηση ε, θα πρέπει να υπάρχει πλαισίωση ιατρική οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πάντοτε υπάρχουν ιατρικοί κίνδυνοι σε κάθε οικίηση πολλές φορές διακυβεύεται η ίδια η ζωή ε, οπότε θα πρέπει να καλύψουμε μια γυναίκα που είναι μόνη της, θα πρέπει να την ε, ενημερώσουμε, να ξέρει τι ισχύει όσον αφορά τις οικίσεις. Ε, Αυτό είναι πρόβλημα εδώ και δεκαετίες. Ε, υπάρχουν τις διακρίσεις επίσης εδώ και δεκαετίες, οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ βασικά που θα πρέπει να αναγνωριστούν, θα πρέπει να αναγνωριστούν ως ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι το δικαίωμα στην υγεία για τις γυναίκες. Είναι θέμα αυτοκαθορισμού, είναι ε, ανθρώπινο δικαίωμα και είχατε αυτό το κείμενο της 12ης ε, Σεπτεμβρίου κατά των, ε, ε, των, των βιαίων, των εξαναγκαστικών και ίσιων. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Και για μας πήγε θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να αποποινικοποιηθεί το δικαίωμα στην διακοπή της κοίησης και θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των σχετικών πολιτικών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πιεστούν τόσο ώστε να ευθυγραμμιστούν με ε, τις πιο προχωρημένες χώρες στην Ένωση που δυστυχώ είναι λίγες. Επίσης έχουμε απαγόρευση πλήρη στην ε, Μάλτα, περισμούς μεγάλους στην Ιρλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, οπότε θα πρέπει να νομιμοποιηθεί το δικαίωμα στην άμβλωση και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κάποιες ε, ρήτρε συνείδησης που αφορούν 80% των γιατρών στην ε, Ιταλία αλλά υπάρχουν προβλήματα ε, και ακόμα και εδώ στο Βέλγιο όσον αφορά ε, την εγγραφή στα Μητρώα ε, των ληξιαρχείων εδώ στο Βέλγιο και υπάρχει ο κίνδυνος κάποιων αντιδραστικών κυβερνήσεων ε, που πολλές φορές επιβάλλουν τις πεπιθήσεις τους στο αστικό δίκαιο και εις βάρος των δικαιωμάτων. Ε, ο φορέας μας αυτό θέλει να σας ε, αναδείξει σήμερα, να σας τα εξηγήσει, διότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ε, διαμαρτυρίες και έχουμε την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην 28 Σεπτεμβρίου την 5 στις 6 ώρα θα κάνουμε αυτή εδώ την διαδήλωση για να υπάρξει αποποινικοποίηση της άμπλωσης. Η διακοπή της κοίησης είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα προς τούτο. Θα πρέπει να υπάρχει ισότητα στην πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό. Χρειάζεται επίσης σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην ε, κατάρτιση ε, και ενημέρωση από σε ειδικών όσον αφορά τις τεχνικές διακοπής της κοίησης. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τελευταία μας διεκδίκηση είναι ότι στηριζόμαστε σε εσάς. Εσείς απευθύνετε έκκληση στα κράτη-μέλη να ευθυγραμμιστούν προς τα πάνω όσον αφορά τις ρυθμίσεις για αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα στην ε, υγεία και στον αυτοκαθαρισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους. Έχουμε 10 λεπτά αγαπητοί συνάδελφοι γιατί στις 6 ώρα έχουμε ψηφοφορία. Λοιπόν, να ξεκινήσει η συζήτηση ο κύριο Γκέρ και μετά η κυρία Πετήρ, Μπιόρκ και Μάρτιν. Παρακαλώ. Δύο λεπτά ο καθένα. ε. Τέσσερα λεπτά θέλω εγώ. Σα παρακαλώ γιατί δεν μπορώ αλλιώ. Εδώ πέρα μιλάμε για οικογενειακό προγραμματισμό. Ε, κοιτάξτε, όταν εγώ και η γυναίκα μου γνωριστήκαμε θέλαμε να κάνουμε 7 παιδιά, είχε μια δύσκολη γέννα, αποφασίσαμε να κάνουμε 4 και να υιοθετήσουμε άλλα 3. Εδώ πέρα λοιπόν υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ άντρα και γυναίκας και έγινε οικογενειακός προγραμματισμός. Έχουμε λοιπόν ευτυχισμένα παιδιά ως αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοούμε οικογενειακός προγραμματισμός. Εδώ πέρα όμως έχουμε μία μονομέρεια. Μιλάμε από την IPPF ε, για μεθόδους προφύλαξης, International Planned Parenthood. Ε, η μητρική της είναι η Planned Parenthood of America και εδώ πέρα έχω την εντύπωση πως αυτή η επιχείρηση πλέον γίνεται business. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Δηλαδή έχουμε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο είτε πουλάει εκτρώσεις είτε χάπια. Εν ολίγης. Στην Αφρική έχουμε διάφορες χώρες ε, που υποφέρουν από μεγάλη θνησιμότητα της μητέρας. Ε, έχουμε μεταξύ αυτών και την 121η χώρα, της Χέρα Λεόνε, στην οποία είπαν ότι νομοποιήστε την έκδοση και θα πέσει η θνησιμότητα της μητέρας. Και όμως δεν έγινε αυτό. Στην Αίγυπτο η έκτρωση απαγορεύεται για λόγους θρησκευτικού. Όσον αφορά λοιπόν τους θανάτου μητέρα, βρίσκεται στην 63η θέση παγκοσμίω. Οπότε το να λέμε ότι η έκτρωση είναι η πανάκια για τον οικογενειακό προγραμματισμό είναι νομίζω λάθος. Με συγχωρείτε, είμαι άνδρα, συγγνώμη που το λέω σε αυτή την αίθουσα, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι προφύλαξης Κατά βάση δηλαδή ε, φτάνει ένα θερμόμετρο. Υπάρχει αυτή η μέθοδος και μπορεί έτσι κάποιος να διαπιστώσει ποιες είναι οι πέντε γόνιμες μέρες του μήνα. Ε, δηλαδή αν επικεντρωθούμε σε αυτό, να το μάθουμε αυτό στις γυναίκες. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα όμως, πρέπει να μπει και ο άντρας κάπου στη διαδικασία. Ε, έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε πράγματα χωρίς χημικές ουσίες. Ε, μιλάμε όμως τώρα για ένα μέσο προφύλαξης, το χάπι. Το AIDS δεν θα ελεγχθεί στην Αφρική και δεν τα καταφέρνουμε γιατί είναι πολύ ακριβά τα μέσα. Και τώρα θέμε στην Αφρική κιόλας να πουλήσουμε αντισυλληπτικά χάπια. Καλύτερο είναι δηλαδή να χτίσουμε νοσοκομεία να μειωθούν οι θάνατοι στη γέννα και κατόπιν να έχουμε έναν αποτελεσματικό οικογενειακό προγραμματισμό ο οποίος ε, δεν θα προσανατολίζεται μόνο στην έκτρωση αλλά θα βρει και άλλους ε, τρόπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Now, Mr. Κυρία Πετήρ, σας παρακαλώ ε, σύντομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έγιναν λανθασμένες ε, δηλώσεις. Ε, το αγέννητο παιδί είναι ζωντανό από τη στιγμή της σύλληψης και έχει τα ίδια δικαιώματα όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Η συνεχής πίεση για τις ακτρώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη δεν έχει βάση στο διεθνές δίκαιο και αντίκειται στην αρχή της επικορικότητας. Η συνεχής αυτή πίεση ε, προς τους βουλευτές των κρατών μελών για να επεκταθεί το δικαίωμα της έκτρασης ε, δεν συμφωνεί και με το κείμενο του ICCPR και με τα όσα έχει αποφανθεί το ΕΣΔΑ σε διεθνείς συμβάσεις και στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν υπάρχει καμία βάση για δικαίωμα στην έκτρωση. Η ICCPR ε, στο άρθρο 6 παραγραφό 5 απαγορεύει την ε, ε, εκτέλεση εγγύων γυναικών προς, για, για να προστατευτούν τα συμφέροντα του αγέννητου παιδιού. Και υπάρχει επίσης δικαίωμα στην προγεννητική υγεία του παιδιού και υπάρχουν και διάφοροι κανονισμοί σε κράτη-μέλη που προστατεύουν την υγεία της μητέρας και του αγέννητου παιδιού. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, μια ευρύτατη ελευθερία για να αξιολογήσουν το πώς θα προστατεύσουν την αγέννητη ζωή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ότι το αγέννητο παιδί είναι μέλος της ανθρώπινης οικογένειας, είναι άνθρωπος χώρες ε, που νομίμως ε, και νομικώς προστατεύουν το αγέννητο παιδί δεν υπονομεύουν την προστασία της υγείας της μητέρας. Χρειάζεται λοιπόν να επισημάνουμε ότι εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πάνε προς την εκπαίδευση των γυναικών σε τρίτες χώρες για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους ε, και τα λοιπά και όχι να τους μαθαίνουμε για την αντισύλληψη. Εγώ δεν θέλω τα λεφτά μου να χρησιμοποιούνται για αυτό τον στόχο. Γιατί δεν βοηθάμε τα εκατομμύρια γυναίκες που θέλουν ε, να κάνουν κάτι και δεν μπορούν. Για να τελειώσουμε, εγώ θέλω τα λεφτά να πάνε στα αντισυλληπτικά και στις εκτρώσεις ε, και θεωρώ πως η αύξηση των 20 εκατομμυρίων ε, είναι ψίχουλα σε σχέση με τις ανάγκες που αναφέρθηκαν και είχαμε τροπολογίες στην Επιτροπή μας που θα είναι πολύ περισσότερα λεφτά αλλά δυστυχώς κατέψαν με ισχνή πλειοψηφία και θέλω να πω συναδελφούς στην επόμενη ψηφοφορία του χρόνου η Επιτροπή μας να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο να μπει ένα πολύ ψηλότερο ποσό σε αυτές τις γραμμές και ελπίζω να μπορέσουμε να συντονίσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις εντός τη γιατί εάν δεν πάρουμε τα λεφτά η δική μας επιτροπή δεν θα το κάνει καμία άλλη επιτροπή ε, χαιρετίζουν την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ για τα 20 εκατομμύρια αλλά όπως λένε και οι συνάδελφοι από το πάνελ θέλουμε πολύ πολύ περισσότερα λεφτά Έχετε βεβαίως ε, στήριξη στην Επιτροπή μας κάποιοι από εμά εμπλεκόμαστε και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο για τα δικαιώματα αυτά. Προσωπικά εγώ είμαι από τη Σουηδία, θεωρώ ότι η σχέση με την ενδυνάμωση των γυναικών και είναι και ζήτημα το εξής. Αν οι γυναίκες δεν τα καταφέρουν θα είναι πιο ευπαθείς οι γυναίκες και τα κορίτσια και θα έχουμε ε, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που είναι βασανιστήριο. Είναι βία κατά των γυναικών, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είμαστε στο 2017 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των γυναικών ε, και των κοριτσιών και πράγματι αντιμετωπίζουμε αντίσταση αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο εμείς είμαστε ισχυρότεροι και ειδικά οι νέοι ε, θέλουν να βρούμε λύσεις και θα βρούμε Σας ευχαριστώ κυρία Βιόρκ κύριε Μάρτεν Ευχαριστώ πρόεδρε ένιωθα μηχανία, νευρικότητα πριν έρθω εδώ. Γιατί τελικά συζητούμε από μία μεριά το, οι δημοκράτες και από την άλλη μεριά απέναντι είναι οι συντηρητικοί. Μα τι να κάνουμε, να απαγορεύσουμε την αυτοκανοποίηση στους άντρες τόσο ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενεργείας γιατί και εμείς θα πρέπει να δούμε το πώς δεν θα υπάρχουν τα όπλα για να μην γίνεται πόλεμος. Όμως έτσι με αυτά που γίνονται, γιατί με τον πόλεμο εδώ έχουμε πολύ περισσότερα θύματα από όσα από τις αμβλώσεις. Αλλά για πέστε μου, τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία της Σουηδίας, κατοχωρών, Δανίας, Βελγίου, ούτως ώστε να αποζημιώνονται οι ΜΚΟ από τις αποφάσεις Τραμπ θα πρέπει να γίνεται εδώ αυθεντική συζήτηση θα πρέπει να μπορούμε να αναλάβουμε τον ρόλο μας θα πρέπει να πιέζουμε τα κρατημέλη θα πρέπει να υπάρχει όντως αυτή η ε, αποζημίωση γιατί οι γυναίκες στην Ευρώπη και παντού να μπορούν να έχουν αντισυλληπτικά να μου πει, να μου απαντήσει η Κομισιόν τι κάνετε για αυτό Έχετε αναλάβει διαβήματα. Ευχαριστούμε, κυρία Μίλλερ. Πρώτα-πρώτα και εγώ να έρθω να συμφωνήσω με την ε, συνάδελφο Μπιόρκ. Και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για την αντισύλληψη με πάντα τρόπο. Για όλους τους μέθοδους αντισύλληψης. Είναι εφιάλιστο να είναι κανεί έγκυο χωρί να το θέλει. Πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τους βιώσιμους στόχους της ανάπτυξης εδώ είναι και το θέμα τη αντισύλληψη. Έχω παραστεί σε ε, κάποια συνάντηση στα πλαίσια του ΟΗΕ και υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ των όπω γνωρίζουμε. Και σα ερωτώ, σκοπεύετε να χαράξετε μια πιο συνεπή στρατηγική και τι γίνεται το πρόγραμμα δράσης για την εμπραγωγική υγεία του ΠΟΗ που αφορά και την Ευρώπη για το 17 και πέρα. Πρόεδρε, βλέπετε πως η συζήτηση μας είναι απόδειξη του ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει αντίδραση και εδώ στο Κοινοβούλιο. Δίνουμε τη μαγείτη τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ. Οπότε δεν πρόκειται να καμφθούμε από τους αντιθέτους. Δεν λέμε για την αντισύλληψη, λέμε για την γενικό προγραμματισμό, για τα γενετήσια δικαιώματα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως θα υπάρξει η κατάλληλη πρικοδότηση που χρειάζεται. Ο μεγαλύτερος δωρητής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αντισύλληψη βοήθεια. Άρα κάνουμε μια προσπαθιούλα παραπάνω γιατί όσα κάνουμε επηρεάζουν τη ζωή πάρα πολλών γυναικών. Και υπάρχει πρόβλημα τη χρηματοδότηση τώρα. Δεν βλέπουμε να τι ερωτήσει. Επομένω, παρακαλώ να δοθούν οι απαντήσει από του προσκεκλημένου. Παρακαλώ να περιοριστείτε μάξιμουμ στα δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Εκπρόσωπο τη Ντεύκο. Ε, δύσκολο αυτό. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ οικογενειακού προγραμματισμού και έκτρωσης. Δεν είναι το ίδιο. Το ένα γίνεται για να προλάβουμε το άλλο. Η Κομισιόν στηρίζει προγράμματα που έχουν στόχο να βελτιωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός και άρα έτσι προλαμβάνουμε τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και δεν υπάρχει ανάγκη έκτρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προωθεί την έκτρωση ως μέσο οικογενειακού προγραμματισμού. Από την άλλη, σύμφωνα με την Διεθνή ε, Διάσκεψη για τον Πλησμό και την Ανάπτυξη, δεν κάνει διάκριση κατά τέτοιων παρόχων σε χώρες όπου η έκτρωση είναι νόμιμη. Στηρίζουμε λοιπόν τέτοια προγράμματα για να είναι ασφαλής όπου είναι νόμιμη η έκτωση. 200.000 γυναίκες ε, εξακολουθούν να πεθαίνουν στη γέννα ή από εκτρώσεις οι οποίες δεν είναι ασφαλείς ε, ή από περιπλοκές ε, της εγκυμοσύνης. Για τα θέματα τώρα, για το ερώτημα και αν υπάρχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση Νομίζω πως η συζήτηση με τα κράτη-μέλη αντικατοπτρίζει και τι απόψει που ακούστηκαν εδώ πέρα. Υπάρχει όμως συνένεση για το σχέδιο δράσης ε, που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη και που έχει γίνει μέρος του κεκτημένου που εφαρμόζουμε και που σαφώς υπερασπίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα κάθε γυναίκα να αποφασίζει ελεύθερα για την αναπαραγωγική της υγεία. Τώρα, αν ζητάμε περισσότερα κονδύλια προς τα κράτη-μέλη, αυτό νομίζω είναι δουλειά των κρατών μελών, πώς θα χρηματοδοτηθεί η αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά όπως είχα εγώ πει στις αρχικές μου παρατηρήσεις, εξετάζουμε όλα τα προγράμματα, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό. Κύριε Ντενεκερ, να θα είμαι σύντομη. Όπως αναφέρθηκε, το πρόγραμμα δράσης υιοθετήθηκε το 1994 και είναι η βασική μας αρχή θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και να τονίσω και πάλι ότι η πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό μπορεί να μειώσει κατά 1 τρίτο την θνησιμότητα της μητέρας και κατά 20% την παιδική θνησιμότητα και συνολικά πρόκειται για σημαντικό μέσο για να μειώσουμε και τα αφροδίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πολύ που είδα τόσο σημαντική ε, στήριξη και για την ισότητα των φίλων αλλά και για τα γενετήσια και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Είναι προφανές ότι χρειάζονται οι γυναίκες την ελευθερία αυτή καθώς και τη δυνατότητα να μπορούν αυτόνομα να αποφασίσουν. Και χάρηκα που άκουσα στην αρχή και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να δούμε και τις ίδιες δεσμεύσεις να λαμβάνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο για το σχέδιο δράσεως που αποτελεί και την βάση, το θεμέλιο και είναι ένα σχέδιο το οποίο έχουν συμφωνήσει όλες οι χώρες μέλη. Με ορισμένες εξαιρέσεις βέβαια που είχαν επιφυλάξεις, αλλά γενικώ αυτό δείχνει μια ευρωπαϊκή συνένεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσείς Σίλια. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές που στήριξαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των γυναικών και απαντώ στις επιφυλάξεις σας με δύο λόγια. Σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας δέχεται ότι η διακοπή του κετού αποτελεί δικαίωμα για την ε, δικαίωμα της γυναίκας. Και επίσης σε ψήφισμό του τον Σεπτέμβριο καταδικάζει την απαγόρευση αυτή το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει κανένα νομοθέτημα το οποίο να ε, διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμούσα να παρέμβω προηγουμένως, αλλά πρόκειται για μια ε, παρατήρηση πιο πολύ διαδικαστική. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη ένα τόσο σημαντικό θέμα και να επιτρέπεται επί 45 λεπτά και περισσότερο στους παρεμβαίνοντες και μόνο 10 λεπτά για τους βουλευτές. Σας παρακαλώ πολύ, σας συγκεντεύω, γιατί για μια ολόκληρη κοινοβουλευτική περίοδο κατήχα τη θέση σας και προσπάθησα πάντοτε να αφήσω επαρκή χρόνο έκφρασης των απόψεων των ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ ε, πολύ και θα παρέμβω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, thank you very much. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στους πανελίστ, σε όλες και όλους που κάθονται εδώ δίπλα μας. Το τελευταίο θέμα της σημερινής διαταξής μας, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι η ψηφοφορία. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοσιονομικά του 2018, όλοι οι τομείς, ή όλα τα τμήματα. Ε, αν έχετε βεβαίω τι ε, κάρτε σα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μπορούμε να αρχίσουμε αμέσω. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Ματέρα. Τροπολογία 5 υπέρ. Ξαναλέει η πρόεδρος, τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές. Σας παρακαλώ επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Α, ίσως βιάστηκα λέει η Ξαναψηφίσουμε, Λοιπόν, Πέρα εγκρίνεται. Α, το σωστό είναι ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Σε δύο τμήματα. Υπε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, <coughs> εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, αυτό απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Υπέρ λέω. Τρίτη φορά υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είμαι βεβαία. Παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, το σχέδιο γνωμοδοτήσεω στο σύνολό του. Ω τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ακολουθεί. έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια αλλαγή, σε μια μάλλον κοινωνία δημοκρατικής ε, αλλαγής. Κυρία Βαλίνα, η συγκεκριά. Τροπολογία 8, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, υπέρ. Κατά, αποχές, παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας παρακαλώ επαλήθευση. Τέλος. Απερίφθη. Τροπολογία 11. ε, μάλλον ε, αρχίζει η ψηφοφορία λέει πρώτος. Με συγχωρείτε διακόπτη. Δικό μου λάθος. Λοιπόν, τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 με προφορική τροπολογία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αχ, τι έπαθα λέει η πρόεδρος. Υπέρ θέλω να πω, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεκατρία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαναληφθεί αυτή η ψηφοφορία. Πρώτο λοιπόν, ή μάλλον δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, επαλήθευση. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ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 Πέραση της ψήφου. Απερίφθη. 29. Σε πέντε θυμάτα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει ψήφο, η ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ. Ο κύριος Βος, στη δική μας ε, λίστα ψηφοφορίας υπάρχει μια τροπολογία γλωσσικού χαρακτήρα. Και αυτή ήταν το πρώτο τμήμα. Α, ναι, ναι, λέει η πρόεδρος. Θέλετε να ξαναψηφίσουμε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. δεν αναφέρατε την γλωσσικού χαρακτήρα τροπολογία. Την ψηφίσαμε εμείς ως πρώτο τμήμα. No. So we need to. No. Uh, uh, uh, colleagues, we don't δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την γλωσσική τροπολογία. Υπάρχει ένα πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε αυτό το πρώτο τμήμα. Νομίζω τότε κάποιο λάθος κάναμε εμείς, λέει ο κύριος Βός. Να επαναλάβουμε. Καλά. Ωραία. Τροπολογία 29. Πρώτο τμήμα, όχι η γλωσσική τροπολογία. Μόνο το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα λοιπόν ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Καλώς, επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Πέρας. Όντως εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Παρακαλώ επαλήθευση. Αρχίζει η ψήφος, τέλος, απερίφθη. Πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Υπέρ λέω πάλι, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρία σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα Τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τσεκ, ωραία, παρήθευση λοιπόν. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 6, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό ή και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ και τους συζητητές και σκιώδεις εισηγητές, εισηγήτριες. Η επόμενη συνάντησή μας, μην την ξεχάσετε, 10 Οκτωβρίου, 10 Δεκάτου από τις 9 το πρωί και όλη την ημέρα, 10 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ όλα τα μέλη, συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, καθώς και τους μεταφραστές και οι οποίοι ανταποδίδουν. Γεια σας και καλό βράδυ.